τους σωστούς φόρους, να σώζουμε ανθρώπους στη θάλασσα, να προ... μην προωθούμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής που κάνει τα στραβά μάτια όταν πνίγεται κόσμο στη Μεσόγειο. Τέλος, ο πλανήτης χρειάζεται ε, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες για να βγουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι από τη φτώχεια. Το πρόγραμμα ε, μάσας θα πρέπει ε, να ανανεωθεί για να φέρει αποτέλεσμα εμείς ως Γκουε, κυρία Βαντερλάιν, δεν είμαστε έτοιμοι να σας εμπιστευτούμε την Ευρώπη. Ο κόσμος και ο πλανήτης χρειάζεται καλύτερο. Ευχαριστούμε ο κύριος Λιγκούτκο. Και εσείς δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή σας αποτελεί την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα και ελπίζουμε όντως να πρόκειται για ένα νέο ξεκίνημα. Η ομάδα μας σας στηρίζει για πολλά πράγματα. Σίγουρα σας στηρίζουμε για, να, για την επιτυχία του συμβιβασμού στον προπολογισμό, για την ενιαία αγορά που ανοίγει και στις υπηρεσίες για να βρεθούν λύσεις όσον αφορά το μεταναστευτικό, για την εφαρμογή ε, μέτρων φιλόδοξων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά πρέπει να τονίσω ότι εμεί θα στηρίξουμε και τις κοινότητες των οποίων η ζωή απειλείται από τις υπερβολικές μερικές φορές κλιματικές φιλοδοξίες. Να έχετε υπόψη σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 26-28 κυρίαρχες χώρες και όλες οι χώρες μετράνε εξίσου. Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε εξουσίες από τις χώρες μέλη, ε, προθώντας ε, την αρνησικυρία, τα βέτο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι που θέτει τους στόχους της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης πάντως και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε σας παρακαλώ μην συνεχίζετε τις πρακτικές που εφάρμοζε και η προηγούμενη Επιτροπή που τελικά παραβίαζε και το πνεύμα και το γράμμα των συνθήκων όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Παρόλα αυτά που ακούτε εδώ στο ημικύκλιο αυτό ή στις διάφορες αίθουσες της ε, Βρυξέλλες, δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, σας παρακαλώ, να εφαρμόσετε μια πολιτική που να βασίζεται σε δεδομένα και σε στοιχεία και όχι τα δεδομένα και τα στοιχεία να βασίζονται σε πολιτικές. Ευχαριστούμε κύριο Τζάνι. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε Βαντερλάιν, επιτέλους μετά από μήνες διαφωνιών ε, μεταξύ των διαφόρων μερών που συνθέτουν αυτή την πλειοψηφία. Έχουμε μια επιτροπή δυστυχώ σε εποχέ μεγάλη κρίση, τι μεγαλύτερε που βιώνουν ποτέ τα ευρωπαϊκά όργανα και θα έχουμε έτσι ξαφνικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι η πιο αδύναμη που είδαμε ποτέ, που ήδη κουτσένει και που βάσει των όσων λέτε εσεί και των υποσχέσεών σα το τελευταίο εξάμεινο φαίνεται να είναι και τυφλή. Δεν ε, έχει καταλάβει το μήνυμα που στέλνουν οι Ευρωπαίοι πολίτε και αρνείται να προτείνει μια ε, ρηξικέλευτη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες μας. Εσείς στην ομιλία σας σήμερα αναφερθήκατε σε gender balance, σε green new deal, αλλά δυστυχώς όμως αυτό που, που αισθάνονται το πρωί όταν ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι πολίτες Δεν είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ισορροπημένη από ψηφίλου. Σκέφτεται πώ θα τα βγάλουν πέρα οικονομικά μέχρι το τέλος του μήνα. Πώ θα βρουν δουλειά. Πώ θα καταφέρουν να ζήσουν με τους μισθούς τους, με τους μισθούς που παίρνουν και για την νέα πράσινη συμφωνία φαίνεται να έχετε μια ιδεολογική προσέγγιση. Αυτό δεν θα θέλαμε να οδηγήσει σε περαιτέρω ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις δικές μας επιχειρήσεις. Η Ευρώπη ήδη έχει κάνει πολλά ε, για τη μείωση των εκπομπών. Άλλοι εκτό Ευρώπη πρέπει να κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν μπορούν οι δικέ σα διατάξει και τα δικά σα νομοθετήματα για αυτό το θέμα να αποτελέσουν επιπλέον βάρο και για τι οικονομίε και για τι επιχειρήσει μα δεν άκουσα να μιλάτε για θέματα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν απειλές προς την ανταγωνιστικότητά μας ε, εκ των έξω, αλλά δεν μας προτείνετε να διορθώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής μας αγοράς. Δεν μιλάτε για το κοινωνικό ντάμπινγκ, για το μισθολογικό ντάμπινγκ που λαμβάνει η χώρα εντός της Ένωσης. Δεν άκουσα να λέτε τίποτα για το φορολογικό ντάμπινγκ και για την αποβιομηχανοποίηση που αυτή τη στιγμή ε, συντελούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταστρέφουν την εσωτερική μας αγορά με περηφάνεια η ομάδα μας σήμερα θα πει όχι σε ανθρώπου σαν εσά που με την αδράνειά σα θέλετε πραγματικά να καταστρέψετε την Ευρώπη. Εγώ σα προτείνω, αμφισβητήστε του εαυτού σα, καταλάβετε τι λάθη έχετε κάνει με τι πολιτικέ που έχετε προωθήσει στο παρελθόν και αλλάξτε πορεία βάσει των επιθυμιών των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλιώ η Ευρώπη δυστυχώ δεν πρόκειται να έχει μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Κέλλερ, δύο λεπτά, ε, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αναλαμβάνει. Είναι επιτροπή όταν η κλιματική αλλαγή μας δείχνει ότι δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε και ότι όντω αποτελούν προτεραιότητα, όπως αποτελούν προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για το 90% των Ευρωπαίων. Όμως παρόλα αυτά δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτοί οι τίτλοι θα προχωρήσουν και σε δράση γιατί δεν αλλάζει η πολιτική, η γεωργική, η εμπορική, οπότε τα κλιματικά μέτρα θα μείνουν στη μέση. Βέβαια χαιρόμαστε ότι έχουμε περισσότερες γυναίκες από ποτέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες κυβερνήσεις τελικά μπορούν να βρουν γυναίκες. Άρα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά για να επιτευχθεί ισορροπή μεταξύ των δύο φίλων και καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην κοινωνία γενικότερα. Ακούσαμε ε, ότι υπάρχουν πολύ καλοί υποψήφοι, πράγματι, αλλά υπάρχουν και μερικοί που μα βάζουν πολλέ αμφιβολίε. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι σοβαροί όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ αξίε. Κυρία Πρόεδρε, ε, δεν θα υποστηρίξουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν είναι σαφή για αυτά τα πράγματα. Κάθε φορά που αναλαμβάνεται μια πρωτοβουλία πάντω που προστατεύει το περιβάλλον, που ενισχύει την κοινωνική Ευρώπη, που ενισχύει το κράτο δικαίου, είμαστε έτοιμοι να σα στηρίξουμε αλλά θα το λέμε επίση κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάτι στραβό ή δεν κάνει αρκετά. Η Ευρώπη πρέπει να είναι αποφασιστική τώρα και ελπίζω να καταλάβετε ότι χρειάζεται θάρρο και να έχετε τη δύναμη να υψώσετε το ανάστημά σα απέναντι στο Συμβούλιο όταν δεν θέλει να ακολουθήσει, όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, όταν πρόκειται για κράτο δικαίου. Εμεί θέλουμε τη δράση, γιατί πρέπει να αναλυφθεί η δράση τώρα. Ε, γι' αυτό δεν σα δίνουμε κόκκινη κάρτα, παρόλο που υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερα και τα έχουμε πει και ξαναπεί πολλές φορές και δεν βλέπουμε να ανταποκρίνεστε. Αλλά δεν θέλουμε να σας δώσουμε ούτε και λευκή επιταγή και γι' αυτό αποφάσισε η ομάδα μας να κρατήσει θέση αποχής και να ελπίσει ότι δεν θα διαψεύσετε τις όποιες ελπίδες έχουμε από σας. Σας χρειάζεται σίγουρα θάρρος και ενέργεια όχι απλώς για να διατηρηθεί η Ήπειρος ε, μαζί και ενωμένη, αλλά και για να προωθήσει τις αξίες της. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Πρόεδρε, υπάρχουν πολλά θέματα πάνω στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποδείξει την αποφασιστικότητά της και την αποτελεσματικότητά της για να εξυπηρετήσει τους πολίτες που πιστεύουν στα προγράμματα αυτά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ποτέ δεν είχε η Ευρωπαϊκή, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μια επιτροπή τόσο φιλόδοξη στον τομέα του περιβάλλοντος και του ψηφιακού κόσμου και επίσης στον τομέα της ισότητας των φύλων που είναι σημαντική για όλους. Θα πρέπει να έχουν όλοι την δυνατότητα ισότιμα να εκφραστούν να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου, να προστατεύσουμε τις ατομικές ελευθερίες. Ποτέ δεν κάναμε τόσο εξαντλητικό διάλογο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ σφράγισε τις πολιτικές αυτές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομάδα μας θα στηρίξει την Επιτροπή σας, αλλά δεν σας δίνουμε επιταγή λευκή. Όσοι θεωρούν ότι η ισότητα και το κράτος δικαίου και το περιβάλλον έχουν ε, σαν λάβαρο, περιμένουν πράξεις και όχι μόνο ευχές και λόγια. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια τίμια και ειλικρινή ε, εταιρική σχέση. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, ε, δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα και τότε το Renew δεν θα σας στηρίζει πλέον. Κάθε επίτροπος έχει ένα συγκεκριμένο ε, ρόλο να παίξει έτσι ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να αγαπήσει πάλι την Ευρώπη. Από το βορρά στο νότο και από την Ανατολή στη Δύση θέλουμε να ξανακάνουμε ελκυστικό και άξιο ε, την ευρωπαϊκή προοπτική. Θέλουμε αυτό να το κάνουμε όχι με λόγια αλλά με γεγονότα που καθιστούν χρήσιμη και ελκυστική την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινότητα του πολίτη. Ευχαριστώ και εσείς τώρα δύο λεπτά κυρία Γκαρθία Πέρες, κυρία Γκαρθία Πέρες. Ευχαριστώ. Τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πέρυσι πιο συγκεκριμένα οι Ευρωπαίοι πολίτες μας έδειξαν ότι θέλουν μια Ευρώπη που να αποτελεί ένα χώρο ευκαιριών. Η σοσιαλιστική ομάδα είναι ξεκάθαρη για το τι πρέπει να κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα εργαστούμε λοιπόν για μια περισσότερο οικολογική Ευρώπη. Για μια Ευρώπη που να είναι περισσότερο φεμινιστική, περισσότερο κοινωνική. Και ελπίζουμε και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει υπεύθυνα. Ελπίζουμε να δράσει με θάρρος θα σας επιτρέψουμε ακόμα και να κάνετε λάθος, αλλά δεν θα σας επιτρέψουμε ποτέ να παρετηθείτε, να μείνετε σε αδράνεια, να μην είσαστε ικανοί να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στο μέλλον. Θα είμαστε λοιπόν σε επιφυλακή. Θα παρακολουθούμε, θα συνεργαστούμε, θα ελέγχουμε και είμαι σίγουρη ότι έχουμε μπροστά μας πέντε χρόνια εντατικής δουλειάς για να αποκατασταθεί η ελπίδα στους Ευρωπαίους που πιστεύουν σε διάφορα πράγματα τα οποία περιμένουν και να ελοπιθούν από εσά στο μέλλον. Ευχαριστούμε, κύριο Σβέμπερ. Δύο λεπτά επίση. Κυρία Πρόεδρε, ζούμε σε εποχέ όπου είναι δημοφιλέ ε, και στα μέσα κοινωνική δικτύωση ακραίε θέσει. Αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει σήμερα η παρουσίαση της κυρίας Βάντερ Λάιεν, να καθησυχάσει τα πνεύματα, ε, να συνεργαστούμε από κοινού για την Ήπειρο μας. Σήμερα ε, παρουσιαστήκατε με σθένος ε, ε, για να αναλάβετε αυτή τη δημοκρατική εντολή. Οι επίτροποι προτάθηκαν μέσω του Συμβουλίου από τα κράτη-μέλη αλλά θα συνεργαστούν μαζί με το Κοινοβούλιο. Εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και εμεί εκφράσαμε την υποστήριξή μα προ αυτού. Όλοι το Κοινοβούλιο και οι Κομισιόν θα πρέπει να δημιουργήσουν μια εταιρική σχέση για να συνεργαστούν για την Ευρώπη. Αυτή την ευθύνη έχουμε. Και τώρα εδώ ακούω συμπεράσματα από την αριστερά και δυστυχώς από πολλούς ε, δεξιούς ε, σε αυτό το κοινοβούλιο ε, να μιλούν με τέτοια επιθετικότητα προς την Κομισιόν. Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Είναι η καλύτερη Κομισιόν που μπορούμε να έχουμε για να αρχίσουμε να φέρνουμε αποτελέσματα. Let's start to deliver. Let's start to deliver strong and united European Union. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στις ψηφοφορίες να σας ενημερώσω ότι εκτάκτως ε, οι επεξηγήσεις ψήφου θα γίνουν αύριο αλλά μπορούν να κατατεθούν και γραπτός εφόσον το επιθυμείτε. Με βάση λοιπόν το άρθρο 125 του κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκλέγει ή απορρίπτει με την πλειοψηφία των ψήφων που είναι, των βουλευτών που είναι παρόντες. Μόλις ε, λήξει η ψηφοφορία, εγώ θα υπογράψω την επιστολή ε, διακίνωσης του αποτελέσματος και θα ενημερώσω μέσω αυτής επίσημα το Συμβούλιο. Επ' αυτής της βάσεως θα ε, διορίσει επίσημα με τη σειρά του πάλι το Συμβούλιο την συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Hanno votato tutti? Ψήφισαν άπαντες, τη ψηφοφορίας. Approvato. 461 voti favorevoli. 461 υπέρ, 157 κοτά, 89 αποχές.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 Παρακαλώ καθίστε πρόεδρε. Πριν ε, υπογράψω λοιπόν την πράξη διορισμού θα ήθελα να πω στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι είμαστε υπερήφανοι για τον ρόλο που έπαιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολουθήθηκε μια σοβαρή, διαφανής και δημοκρατική διαδικασία η οποία σεβάστηκε τις συνθήκες και τον κανονισμό. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, τους προέδρους τους, όλους τους βουλευτές και όλες τις πολιτικές ομάδες. Να υπογραμμίσω την πολύ σοβαρή δουλειά που έκανε και η διοίκηση του Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα ενημέρωσης και τον τύπο για την προσοχή τους που έστρεψαν προς τις εργασίες μας. Στρέφομαι τώρα προς την νέα πρόεδρο και της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Υπογράφω τώρα την επιστολή. Και θα πρέπει να την παραδώσω, λέει ο Πρόεδρος. Eh, Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την σημερινή ημερήσια διάταξη. Έχουμε κάποιες σημαντικές ψηφοφορίες μπροστά μας. Έχουμε καταρχάς την έκθεση Καϊλή, κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα. Μία η ψηφοφορία ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τη της ψηφοφορίας. Δεκτή η πρόταση. Τώρα έκθεση Χόλμαϊερ για τον μηχανισμό ευελιξίας. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Δεύτερη έκθεση Χολμάγερ, κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή η πρόταση. Έκθεση επίσης τρίτη Χολτμάιερ και Γκουάντια Σάβαλ για τη διαδικασία προϋπολογισμού για το 2020 κοινό σχέδιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Θέλει το λόγο το Συμβούλιο. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμοι προβλεφτές, κυρίες και κύριοι, σας συγχαίρω που ολοκληρώσατε ε, το έργο σας όσον αφορά την απόφαση για το προπολογισμό για το 2020. Το Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμφώνησε στις 18 Νοεμβρίου στην συνδρίαση συνδιαλλαγής με μεγάλη πολιτική στήριξη. Και υποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Γιώχαν Φανόβερφελτ, τον πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών και του ηγητέ Μόνικα Χολχάγερε και την ε, κυρία Μπαστασαμπάλ, όπω επίση και του υπόλοιπου ευρωβουλευτέ που συμμετείχαν στην δημοσιονομική αυτή διαδικασία για την επικοδομητική του προσέγγιση. Θέλω επίσης να ευχαριστώ και τον Επίτροπο σας ευχαριστώ. Το κοινό σχέδιο ε, επί του οποίου επέτυχε συμφωνία στις 18 Νοεμβρίου το, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο η δημοσιονομική διαδικασία εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 314 ε, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία για τον προϋπολογισμό λοιπόν του 2020 μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Δηλώνω λοιπόν ότι οριστικά εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 και θα προβώ τώρα στην υπογραφή του προϋπολογισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, να στέλνετε η συνεδρίαση για λίγα λεπτά. Και ευχαριστώ για τη συνεργασία σας ε, αυτό το πολύ σημαντικό πρωινό.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 Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Περνάμε στην τελετή απονομής του βραβείου Λούξ. Παρακαλώ να καθίσουν οι συνάδελφοι. Mr. President, ladies and gentlemen. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι υποψηφιώτες για το βραβείο Λουξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το Cold Case Hammersholt. God exists, her name is Petrunia και The Realm. Παρακαλούμε, καλώς ορίστε. Τον ε, σκηνοθέτη Μάτσα Μπρούγκερ και τον ε, παραγωγό της ταινίας ε, Cold Case Hammerheld. Representing the North Macedonian, Belgian, Slovenian εκ μέρου ε, τη συμπαραγωγή Βόρεια Μακεδονία, Βελγίου, Σλοβενία, Γαλλία, Κροατία, ο Θεός υπάρχει, το όνομά του είναι Πετρούνια, η σκηνοθέτης και η παραγωγή. representing και εκπρόσωποι της γαλλο-ισπανικής συμπαραγωγής, ο Αντώνιο Ντελατόρε, ο ε, ηθοποιός ε, του, της ταινίας ε, «Ο και ο παραγωγός. Τώρα ο πρόεδρος θα απονείμει το βραβείο Λουξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2019. Αγαπητοί σκηνοθέτε, ε, κυρία Επίτροπε, Αντιπρόεδρε Ντόμπρεβ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κινηματογράφος είναι ένα κλειδί που ανοίγει τις πόρτες της κατανόησης της πραγματικότητας μας. Βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα ποιοι είμαστε. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος ανέκαθεν περιγράφει λεπτομερώς τις πολύπλοκες κοινωνίες μας, που μερικές φορές είναι δυσνόητες.